Tisztelt képviselőtársaim, Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Παίρνουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τις δηλώσεις της ΥΠΑ της εκπροσώπου ε, για την εξωτερική πολιτική και Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση στην Τουρκία. Παρακαλώ την κυρία Μογκερίνη να λάβει το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε Μογκερίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.